Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, μου ανακοινώνουν ότι βρίσκονται στο διάδρομο ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Σεύκοβιτς, καθώς επίσης και ο κύριος Ραπκάη, που είναι εισηγητής. Όχι, νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να διακόψουμε. Ένα λεπτό ας περιμένουμε γιατί ήρθα και εγώ τρέχοντας από την ίδια συνεδρίαση που συμμετείχαν και εκείνοι, αλλά από ό,τι φαίνεται εκείνοι έρχονται με το πάσο τους και όχι με βήμα γοργό που ήρθα εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάιερ που είναι παρόν και να το παρακαλέσω να δείξει λίγη υπομονή, ένα λεπτάκι μέχρι να καταφτάσουν και οι υπόλοιποι και ιδιαίτερα επίτροπο. In any case, Gay, we don't listen to you because you don't have the microphone. We're going to. Gay Mitchell, δεν σε ακούμε τι λες, γιατί δεν έχεις μικρόφωνο. Σε δέκα δεύτερα αρχίζουμε, λέει ο πρόεδρος τον κύριο Μίτσελ. No, entonces vamos a, vamos a empezar el debate. Ε, ας αρχίσουμε λοιπόν και ελπίζω να καταφτάσουν και οι υπόλοιποι. Γιατί μου είπαν ότι είναι καθοδόν και ο κύριο Ζαπκά. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται η συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ήρθατε και εσεί τρέχοντας. Και εγώ τρέχοντα ήρθα. Αλλά έφτασα λίγα λεπτά νωρίτερα. Το επόμενο θέμα γνωρίζετε ότι είναι η έκθεση του νοέφου Σάγερ, έλεγχο από τα κράτη-μέλη τη άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο καταρχά στον εισηγητή μα, τον κύριο Σάγερ για τέσσερα λεπτά. Γνωρίζετε ότι ε, μπορείτε να μιλήσετε στη συνέχεια και άλλα δύο λεπτά και αν μιλήσετε πάνω από τέσσερα λεπτά τώρα θα σας ειδοποιήσουμε αλλά θα σας αφαιρεθεί ο χρόνος από την τελική σας ε, τοποθέτηση από τη δευτερολογία σας. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας, στην οποία προβλέπονται σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο κοινοβούλιο μας έχουμε ήδη συζητήσει πριν από μερικούς μήνες τη δική μου την έκθεση για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Η κατεξοδότηση πράξη είναι πράξη στην περίπτωση εκείνη που υπάρχει μία μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί όμως η μεταφορά αυτή αρμοδιοτήτων να γίνει και αντίστροφα και μπορούμε σε κάθε περίπτωση να αντιταχθούμε σε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, στο πλαίσιο της υφιστάμενης πρότασης για το άρθρο 291 ε, της συνθήκης μιλάμε για τις εκτελεστικές πράξεις. Στην περίπτωση αυτή τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Εδώ είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία εξασκούν τα δικαιώματά τους για την υλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας. Υπάρχει λοιπόν μια σαφής διάκριση ανάμεσα στις κατεξουδότης πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις. Με την νέα αυτή λοιπόν συνθήκη μας δίνονται πολύ σημαντικές αρμοδιότητες αλλάζει σημαντικά η δυνατότητα επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυξάνουν ουσιαστικά σημαντικά, ιδίω σε συγκεκριμένου τομεί. Όσον αφορά τώρα τι εκτελεστικέ πράξει, έχουμε το δικαίωμα ω νομοθέτη, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ρυθμίζουμε την όλη διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη επιβάλλουν η κοινοτική νομοθεσία στην, στο κράτος τους. Μετά από σημαντικές λοιπόν διαπραγματεύσεις που γίνανε, αποφασίσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θέλουμε να έχουμε σαφή δέσμευση και από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι θα τηρούνται, ότι θα προασπίζονται τα δικαιώματά του. Και μετά από πολύ σημαντικές συζητήσεις καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στον τομέα των εκτελεστικών πράξεων αλλά και στον τομέα των κατεξοδότηση πράξεων. Ακόμα και στην περίπτωση των εκτελεστικών πράξεων καταφέραμε να διατηρήσουμε το δικαίωμα ελέγχου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βάσει της συμφωνίας με, τις, με τα άλλα θεσμικά όργανα προβλέπεται μια συγκεκριμένη διαδικασία που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Η πρώτη σημαντική μου προτεραιότητα ήταν να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την σημαντική μας αυτή θέση. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αναλύσουμε. Υπάρχουν κάποιες ενεξελίξεις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ιδίως στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, καθώς επίσης και στην Επιτροπή Ανάπτυξης, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου γίνονται πολύ σημαντικές συζητήσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα χρηματοδοτικά μέσα και πώς αυτά θα μπορούσαν να ρυθμιστούν. Στόχος μου λοιπόν στο συγκεκριμένο πλαίσιο ήταν ο κανονισμός αυτός να μην προκαταλαμβάνει τη συζήτηση αυτή. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας οι οποίοι δίνουν μάχη σε άλλες επιτροπές αυτή τη στιγμή, στις συζητήσεις δηλαδή που διεξάγουν με το Συμβούλιο και θέλουμε να πετύχουμε βέβαια εν τέλει τη συνεργασία του Συμβουλίου προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ολοκληρώθηκε ο χρόνο μου. Θα ήθελα να πω προ το Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι του ευχαριστώ για την ευελιξία που δείξανε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση και συνειδητοποιώ ότι στο Συμβούλιο ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξετε σε κάποια συμφωνία. Πρόκειται για τη συμφωνία την οποία ήθελε εξ αρχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια συμφωνία που είναι ικανοποιητική για όλα τα μέλη γιατί δεν μιλάμε μόνο για τι συγκεκριμένε πράξεις στα πλαίσια τη συμφωνία αυτή, αλλά περιμένουμε τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το Συμβούλιο να συμμετέχουν στην ε, μελλοντική κοινή συμφωνία που θα προκύψει για τα δύο αυτά σημαντικά ζητήματα, καθώς επίσης και στις δηλώσει που θα γίνουν. Και θέλουμε μια δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ευθυγράμμιση του εναπομείναντος κοινοτικού κεκτημένου. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε και το επιπλέον κείμενο στο εγγραφό μου, το οποίο πιστεύω ότι βρίσκει σύμφωνο όλα τα, όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ναι, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα περίπλοκο. Λοιπόν, να σεβόμαστε απλώ τα χρονικά περιθώρια. Παρακαλώ πολύ. Όμω θα μπορούσαμε να είμαστε και πιο γενναιόδοροι, γιατί είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Πρέπει να εκφράσουμε τα επιχειρήματά μας και να μπορούμε να εκφραστούμε σωστά. Κύριε Πίτρο Πεσεύκοβιτς, έχετε το λόγο. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you very much, Mr. President. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί Είδαμε πάρα πολύ καλές συζητήσεις για την πρωτοβουλία των πολιτών και τώρα ερχόμαστε να συζητήσουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα της επιτροπολογίας. Είναι πολύ καλό σημάδι επίσης ότι μετά τη θέση σε ισχύ της σύνθηκης Λισαβόνας Ολοκληρώνουμε τώρα τα βασικά στοιχεία της νομοθεσίας που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή τους. Ο κανονισμός ε, για τις ελεκτριστικές αρμοδιότητες έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Νόμο στο μέλλον. Θα έχει μεγάλη επιρροή στη δυνατότητα της Ένωσης να κάνει ασκή πολιτική υπέρ των πολιτών της και στο συμφέρον των πολιτών της. Όταν ε, καταθέσαμε την πρόταση, βάλαμε το νέο πλαίσιο για τις εκτελεστικές αρμοδιότητες, πιο απλό, πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές και σε πλήρη εφαρμογή και ε, υλοποίηση της συνθήκης. Ο μηχανισμός που προβλέπεται από τον κανονισμό βασίζεται στην επιτροπολογία, που σημαίνει επιτροπές που να ε, προσωπούν τα κράτη-μέλη, βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέτρα, αλλά δεν θα συμμετέχει το Συμβούλιο αυτό καθ' αυτό, όπως ορίζει η συνθήκη. Μόνο τα κράτη-μέλη και όχι το Συμβούλιο μπορούν να ελέγχουν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες και εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, ο κανονισμός προβλέπει ότι όλες οι ειδικές ε, ε, ρυθμίσεις ε, καταργούνται και ό,τι έχει να κάνει με το anti-dumping και άλλα συναφή θα ε, ρυθμίζονται. Αυτό είναι πραγματική επανάσταση στον τομέα της εμπορικής πολιτικής. Θέλουμε να έχουμε πιο απλές διαδικασίες. Αυτό τι σημαίνει. Όχι μόνο δύο ε, διαδικασίες με το νέο πλαίσιο αλλά και αυτόματη προσαρμογή των σημερινών διαδικασιών επιτροπολογίας και θα αρχίσουν όλα αυτά να ισχύουν για ε, όλη την νομοθεσία από την πρώτη μέρα και αυτό βεβαίως με την επιφύλαξη ε, των εξουσιών που χωρούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλο το κεκτημένο θα ευθυγραμμιστεί με το καθεστώς των κατεξουσιοδότηση ε, πράξεων. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για σας. 153 νομοθετήματα ε, δεν ήταν στη συναπόφαση πριν τη συνθήκη τη Αβώνα και χωρούν αρμοδιότητες τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα γίνουν κατεξουσιοδότηση. Επιπλέον 299 πράξεις ήταν ε, στη διαδικασία που είναι γνωστή ως ΠΡΟΑΚ. Ε, ε, στόχος όμως είναι λήξει η παρούσα κοινοβουλευτική θητεία όλη η νομοθεσία να έχει πλήρως ευθυγραμμιστεί με τις νέες διατάξεις της Συνθήκης Λισαβόνας. Αυτό σημαίνει πλήρη ευθυγράμμιση και ξέρετε πόσο φιλόδοξος είναι αυτός ο στόχος. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερος κύριε Πρόεδρε που ο Βέλγος Υπουργός Σαστέλ είχε την καλοσύνη να μου ζητήσει να δεσμευτώ ενώπιό σα και να δηλώσω και εξ ονόματο τη Προεδρία τα εξή. Η Βελγική Προεδρία γνωρίζει ε, τι φιλόδοξε προθέσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν προκειμένου και καλωσορίζει ε, τι προθέσει αυτέ και υποστηρίζει του στόχου τη. Μπορεί να επιβεβαιώσει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε η ευθυγράμμιση και η προσαρμογή να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Αυτή τη στιγμή υποβληθούν οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πρόθυμη Προεδρία να συνεργαστεί πιστά με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτυχθούν αυτοί οι στόχοι. Και βεβαίω αυτό ε, θέλει να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Ε, και ε, είναι πραγματικά πολύ επικοδομητικό το πνεύμα και συναδελφική η προσέγγιση της Βελγικής Προεδρίας. Θέλουμε ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό, δηλαδή οι νέοι κανόνες να αντικατοπτρίζουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μία εξαίρεση που μας λυπεί και θα επανέλθω στη συνέχεια. Για ποιο λόγο. Μόνο η δική πλειοψηφία μπορεί να εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το να εγκρίνει κάτι. Ποια είναι η εξαίρεση ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θετική γνώμη για ε, μέτρα ε, εξασφάλισης πολυμερών εμπορικών συμφωνιών. Το ξέρουμε ότι είναι περιορισμένο αυτό, αλλά ήμασταν κατά της εξαίρεσης. Θα θέλαμε πλήρη ευθυγράμμιση των πάντων με τους νέους κανόνες, χωρίς εξαιρέσεις. Το λέω αυτό από θεσμικής πλευράς, παρόλο που τελικά ήταν η μόνη βάση για το συμβιβασμό ε, για τον νομοθέτη. Θέλουμε ένα σύστημα πιο διαφανές η όλη διαδικασία θα γίνεται σε πλήρη διαφάνεια. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στις επιτροπές ταυτόχρονα στέλνονται και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Με δικαίωμα ελέγχου, με πλήρη ισότητα και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λένε ότι θεωρεί ενδεχομένω ότι υπερβαίνει τις εξουσίες της και έχετε το δικαίωμα να μας το ε, επισημαίνετε. Κύριε Πρόεδρε, συνοψίζω και τελειώνω. Γνωρίζουμε ότι το κείμενο είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για την Ευρώπη, ενισχύει την κοινοτική μέθοδο σαφέστατα και διευρύνει τις ε, αρμοδιότητες ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, ο νέος κανονισμός προβλέπει ότι σε ορισμένε περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποχρεωθεί να ε, προσφύγει σε μια επιτροπή ε, προσφυγής. Ε, θα είναι όμως μια κανονική επιτροπή και πάλι με ειδική πλειοψηφία μπορεί να καταψηφιστεί το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μην εγκριθεί. Εάν εγκριθεί λοιπόν ο κανονισμός αυτό σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ταχύτατα θα τεθεί σε ισχύ 1η, Τρίτου 2011. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό νέο. Το πλαίσιο αυτό θέλουμε να αρχίσει να λειτουργεί το συντομότερο και ελπίζουμε παράλληλα να ξεκινήσουμε και τα υπόλοιπα και για τις ε, κατεξουσιδότητες πράξεις και για τις εκτελεστικές αρμοδιότητες για να αποφύγουμε ε, τις διαμάχες ε, και ε, τις ε, προστρίβες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σάιε ε, για τη στάση του και το έργο του καθ' όλη τη διαδικασία καθώς επίσης και όλες τις πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία και την ευελιξία που επιδεικνύουν. Και τέλος να ευχαριστήσω τη Βαλγική Προεδρία που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στο Συμβούλιο ε, βρήκε αυτό το τόσο δύσκολο συμβιβασμό και ελπίζω αύριο να εγκρίνετε αυτά που σας προτείνω. Είναι πάρα πολύ καλή υπόθεση αυτή για την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ακολουθούν τώρα οι μιλητές εξ των ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών τους. Πολλούς δεν τους βλέπω. Για παράδειγμα τον κύριο Αλμπερτίνη που κανονικά θα έπρεπε να μιλήσει εξονόμενο τη Επιτροπή Εξωτερικών. Αλλά ευτυχώ παρευρίσκεται ο συνάδελφο Μίτσελ, που θα πάρει το λόγο εξ τη Επιτροπή Ανάπτυξη. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Σάιο, για την προσπάθειά του και την έκθεσή του. Μετά από την έναρξη ισχύω συνθήκη τη Λισαβόνα, ε, η διαδικασία επιτροπολογία θα υποκατασταθεί από τι εκτελεστικέ και τι κατεξιοδόκη πράξει ε, βάσει των άρθρων 290-291, όπω έχει εξηγηθεί. Όμω, εμένα με ανησυχεί ο ρόλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην εφαρμογή των αποφάσεων σε σχέση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Από ό,τι κατάλαβα, είπε μόλι ο Επίτροπο ότι ο στόχο μα είναι μέχρι το τέλο Μέλο τη κοινοβουλευτική θητεία. δηλαδή άλλα 3,5 χρόνια στόχο. Κοιτάξτε, εδώ είναι το κοινοβούλιο, δεν είναι ένα σύλλογο. Αν το συμβούλιο συμμετέχει, το κοινοβούλιο συμμετέχει. Και αυτό. Και πρέπει να πω ως βουλευτής ε, και δεν μου δίνει και ιδιαίτερη χαρά να το πω αυτό ότι φαίνεται ότι μερικές φορές ε, αντί να είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο είναι πολύ κοντά στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο στον όγκο του συχνά πλήττεται από διάσταση απόψεων και μερικές φορές αυτό ε, διευκολύνει την κοινή θέση Συμβουλίου και ε, Επιτροπής κατά τη γνώμη μας. Το Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να ε, πιέζεται να συμφωνήσει απολύτως με τις προτάσεις σε πρώτη ανάγνωση. Το πιο σημαντικό είναι να καταλήξουμε σε ένα δίκαιο συμβιβασμό που θα είναι ο καλύτερος και για το Κοινοβούλιο αλλά και για τους πολίτες που εκπροσωπούμε. Ο κύριος Σάιερ μόλις το είπε, αν αυτό σημαίνει να πάμε σε δεύτερη ανάγνωση, ε, ας πάμε. Αν συμμετέχει το Συμβούλιο, πρέπει να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο κανόνας. Ε, είμαστε συνομοθέτες, υπάρχει συναπόφαση από αυτού. Και ως εισηγητής ε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό Είστε υπερδιπλάσιος, έχετε ξεπεράσει το υπερδιπλάσιο του χρόνου σας. Ήθελα απλώς να πω ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σεβαστεί και το Κοινοβούλιο και δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι αυτός ο συμβιβασμός το επιτυγχάνει αυτό. Ευχαριστώ. Ούτε τον κύριο Βιτάλ Μορέιρα βλέπω που κανονικά θα μιλούσε εξ ονόματος Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου αλλά παρευρίσκεται ο κύριος Ελχαντράουι. Έχει ένα λεπτό για να μας εκθέσει την άποψη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συνάδελφοι, καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Ήταν το θέμα περίπλοκο και πάρα πολύ τεχνικό, όσο και σημαντικό όμω για τι μελλοντικέ μα εργασίε. Για τη δική μα Επιτροπή Μεταφορών η παλιά διαδικασία επιτροπολογίας είχε τέσσερις διαφορετικές δυνατότητες, ήταν πολύ γνωστή για μας και ξέρουμε εδώ και καιρό τι γίνεται με τις εκτελεστικές ε, αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, ο συμβασμός που έχει ε, διαπραγματευτεί ο εισηγητής με το Συμβούλιο μας βρίσκει σύμφωνο. Σε δύο πράγματα θέλω την προσοχή σας παρακαλώ. Πρώτον, όσο γίνεται μεγαλύτερη πληροφόρηση του Κοινοβουλίου και όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου ήδη στο προπαρασκευαστικό στάδιο της λήψης αποφάσεων στην Επιτροπή. Και ένα δεύτερο, θα ήθελα να τονίσω τη μεταβατική περίοδο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θα θέλαμε να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξει στη μετάβαση από το κεκτημένο δηλαδή και την προσαρμογή στη νέα διαδικασία να μην ε, είναι ε, απούσα να δείξει γενοδορία στο Κοινοβούλιο να συνεργαστεί μαζί μας και ε, αναμένουμε την υλοποίηση όλων αυτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο αγαπητέ συνάδελφε. Ευτυχώς βλέπω και την αγαπητή συνάδελφο κυρία Χιούμπνερ που έχει ένα λεπτό για να μας εκθέσει απόψη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Eh, uh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπω ο Γκάι Μίτσελ, έτσι και εγώ ανησυχώ αυτή τη στιγμή με την χρήση που γίνεται για τις ε, εκτελεστικές ε, πράξεις, ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε μια έλλειψη εμπιστοσύνη στη διοργανική συνεργασία. Η ε, πρόταση η οποία έχει γίνει αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να απαιτήσει τη χρησιμοποίηση μέχρι το 2013 τόσο εκτελεστικών πράξεων όσο και κατευθυνότηση πράξεων για την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Νομίζω ότι θα πρέπει σε κατά περίπτωση να αποφασίσουν οι συνομοθέτες ποια από τις δύο μεθόδους θα χρησιμοποιηθεί. Νομίζω ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μοιραστούν τι αρμοδιότητέ του με, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μα περιμένουν δύσκολα χρόνια. Το καθήκον μα ή να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε στο έπαρκο τι πολιτικέ μα και να μην, υπάρχουν... να μην υπάρχει αντιπαράθεση στη διοργανική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ούτε τον κύριο Δεκάστρο βλέπω. Α, τον βλέπω. Ευτυχώ ήρθε ο κύριο Δεκάστρο και θα μας μιλήσει για δύο λεπτά εξ ονόματος Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπέθρου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως επικεφαλής της Επιτροπής Γεωργίας είμαι απογοητευμένος από την έκθεση Ζάιερ την οποία θα ψηφίσουμε αύριο. Καμία από τις τροπολογίες που ομόφωνα στηρίχθηκαν από την Επιτροπή μου και το υπογραμμίζω αυτό δεν ελήφθη υπόψη. Μολονότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι μία από τις ε, πολιτικές εκείνες οι οποίες υπάγονται ιδιαίτερα στην επιτροπολογία και που συμμετέχουν λοιπόν πάρα πολύ στις, ε, στη νέα διαδικασία των εκτελεστικών πράξεων όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνα. Σύμφωνα με το άρθρο 10 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να έχει κανένα περιθώριο διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο όσον αφορά την ε, διαμόρφωση των εκτελεστικών πράξεων για την κοινή γεωργική πολιτική. Ήδη ξέρουμε ότι το Συμβούλιο δεν θέλει να δώσει τη δυνατότητα εκτελεστικών πράξεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίση το Συμβούλιο Συμβούλιο σε καμία περίπτωση δεν θέλει να προωθηθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις γιατί υπάρχει αυτή η αυτόματη προσαρμογή η οποία εξαιρεί τελικά τις εκτελεστικές πράξεις και προβλέπει μόνο κατεξουδότηση πράξης και δεν υπάρχει συγκεκριμένη διορία καταληκτική ημερομηνία γι' αυτό. Επομένως, γι' αυτό το λόγο υπέβαλα με άλλους συναδέλφους μια τροπολογία που ζητώ τουλάχιστον να, να προβλέπετε ένα ενδιάμεσο μεταβατικό μέτρο όσον αφορά την αυτόματη αυτή προσαρμογή. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε σε πρώτη ανάγνωση να, καταφέρουμε, να καταλήξουμε συμφωνία για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο θα καθορίσει τι εργασίε μα τα επόμενα χρόνια. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σημαντικό αυτό ζήτημα να καταφέρουμε να βελτιώσουμε το κείμενο όσο το δυνατόν περισσότερο και να περάσουμε σε δεύτερη ανάγνωση και δεν θα πρέπει να ακούσουμε το Συμβούλιο το οποίο μας απειλεί αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλει να πραγματευτεί εκ νέου την έκθεση αυτή προκειμένου να μας υποχρεώσει τώρα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία πρέπει πραγματικά να τοποθετηθούμε επί του στήματο αυτού, γιατί ουσιαστικά καθορίζει τη διοργανική ισορροπία την οποία θα πρέπει να έχουμε στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε τι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο κλέγεται νόμα και προσωπεί όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Σα ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Πάολο. Το λέω εγώ τώρα, έχει ένα λεπτό συνάδελφο Σάντσες Πρισέδο, εξ ονόμα Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει σημαντικές αλλαγές ε, στην ε, ανάπτυξη και εξέλιξη ε, της ε, νομοθεσίας. Είναι η κατεξουσιοδότηση πράξη και εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ενώ προηγουμένως είχαμε μόνο εκτελεστικά μέτρα. Ο παρόν κανονισμός είναι εκ των όνων κάνευ για να περάσουμε στο νέο σύστημα για τη μετάβαση αυτή και να ε, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκεί ε, τι νέε αρμοδιότητε της σύμφωνα με τι ειδήσει της Λισαβόνα. Ενισχύει τη δημοκρατική αρχή διότι αναγνωρίζει το δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυξάνει τη διαφάνεια με αιτήσια έκθεση και εισάγει και ρήτρα αναθεώρηση για να αξιολογείται αυτό βάσει των εμπειριών που αποκομίζονται. Η Οικονομική Επιτροπή ε, είναι ικανοποιημένη από τα αιτήματα που είχε θέσει. Σε ό,τι αφορά τα χρήματα οικονομικά θα αυξήσει ε, τη νομική ασφάλεια και σε ό,τι αφορά ε, την ε, οδηγία τη λεγόμενη ε, Omnibus, το παλιό σχέδιο αφήνει μια τριετία για να τεθεί σε ισχύ αυτό το νέο σύστημα και ορίζει ε, κάποιον τρόπο για τις τεχνικές προδιαγραφές για την νέα αρχιτεκτονική εποπτεία ε, ε, σε κάθε κλάδο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για να μπορέσουν αυτά να εγκριθούν. Για όλα αυτά λοιπόν ο συντάκτης νομοδότησης Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων αξιολογώ θετικά την έκθεση και τον κύριο Σάιγερ και τον πρόεδρο για την μεγαλοψυχία του. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ Αντωνίν. Ο κύριο Λάινεν απουσιάζει, κύριο Λάινεν, που κανονικά θα μιλούσε εξ ονόματο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, ούτε ο κύριο Γκρέχ παρευρίσκεται. Κανονικά θα μιλούσε εξ ονόματο ε, τη Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών. Ο κύριο Κούν δεν ξέρω αν είναι εδώ. Θα μιλούσε εξ ονόματο τη Επιτροπή Αλία. Δεν του βλέπω. Δεν φαίνεται να είναι παρόντε. Ακολουθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι τώρα εξ ονόματος των πολιτικών τους ομάδων. Και πρώτα απ' όλα ο αγαπητός συνάδελφος κύριος Λένε για δύο λεπτά για να μιλήσει εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι χρειάζονται εδώ κάποιες διευκρινήσεις και στην Ολομέλεια για να διασκεδαστούν οποιασδήποτε αμφιβολίες που ε, ε, ε, προέκυψαν από συζητήσεις στη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών και στις λοιπές συζητήσεις. Περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι ο ορισμός των πράξεων, τι είναι κάτι εξουσιοδότηση πράξης ή τι είναι εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 290 ή 291 της Συνθήκης. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε για την εξουσιοδότηση ε, για το πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα άρθρα. Η διαδικασία λοιπόν, όχι τον ορισμό, σε περίπτωση που ε, εμπίπτει μία περίπτωση στο άρθρο 290-291. Το δεύτερο, κριτική στο άρθρο 10. Και το άρθρο 10 αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία και μόνο, τίποτα άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό εξήγησε και διευκρίνησε ότι βεβαίως έχει την πρόθεση στην εφηγράμμιση όλα τα νομοθετήματα που ισχύουν από την εποχή πριν τη Λισαβόνα να τα ε, προσαρμόσει και να φέρει νέα πρόταση και στους δύο νομοθέτες, και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Αυτό ενισχύθηκε ε, με βάση την προηγούμενη διοργανική συμφωνία. Τι είναι λοιπόν το πραγματικά καινούριο. Ε, είναι ε, το θέμα του προπολογισμού. Βέβαια, ομολογώ ότι η πρόταση συμβασμού της Βελικής Προεδρίας είναι γραφειοκρατική, αλλά είχαμε δύο μειοψηφίες στο Συμβούλιο που μπλόκαραν τα πάντα και θα πρέπει να καταλάβουμε τι, κατάφερε το Συμβούλιο να βγει. Το είπε και ο εισηγητής. Είναι κάτι που δεν προβλέπει η συνθήκη. Ε, είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά και ε, για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και ξεπερνάει και τη συνθήκη. Και νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την έκθεση όπως έχει τώρα χωρίς τροπολογίες και νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε πλέον σε πρώτη ανάγνωση ε, να ε, πετύχουμε περισσότερα, μάλλον σε κάποια, κάποια υποτιθέμενη συνδιαλλαγή αργότερα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω στο έδρανό του τον κύριο Ραπκάη, οπότε και θα δώσουμε το λόγο τώρα στην κυρία Λίχτενμπέργκερ, έξω ονόματος των Πρασίνων. Για 1,5 λεπτό. Αλλά όπω θα διαπιστώσατε, είμαστε πολύ ευέλικτοι με τον χρόνο, κύριε Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ρύθμιση αυτή που μας απασχολεί σήμερα έχει μεγάλη προϊστορία. Σε πολλές επιτροπές είχε πέσει σχεδόν σε αφάνεια. Και τώρα παραμονές του τελικού αποτελέσματος ξύπνησαν κάποιοι συνάδελφοι που δυστυχώς αποσιάζουν από τη σημερινή συζήτηση. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική τους άποψη. Ως πρώην μέλος της συντακτικής συνέλευσης θυμάμαι το πνεύμα της συντακτική συνέλευση, πάρα πολύ έντονο το έχω στο μυαλό μου σε πολλούς τομεί ε, είχε ζητήσει η συνέλευση ξεκάθαρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποκτήσει ορισμένα δικαιώματα και μάλιστα έλεγε ότι όφιλε το Κοινοβούλιο να τα αποκτήσει αυτά για να διαφυλάξει την αξιοπιστία του και στο θεσμικό οικοδόμημα της Ένωσης και στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό λοιπόν που μας ε, πρότεινε η συνέλευση δεν ήταν κάτι το οποίο μας χάρισε κανείς. Χρειάστηκαν πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις και η Βελγική Προεδρία μεσολάβησε στο Συμβούλιο για να γίνουν κάποια σημαντικά βήματα πρόοδου. Θυμίζω αυτό που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος Λένε της μόνιμης δυνατότητας ελέγχου και παρακολούθηση αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπερβαίνει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες. Βέβαια, ορισμένα πράγματα δεν είναι ιδεώδη, όπως οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, αλλά Παρ' όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει μπορώ να συμφωνήσω με το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ τη Βελγική Προεδρία. Πραγματικά κόπιασε πάρα πολύ για να έρθει αυτό σε αίσιο πέρα και κυρίω τον εισηγητή μα που εργάστηκε πάρα πολύ και με το μυαλό και με την καρδιά του. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Οκληρώνονται εδώ οι τοποθετήσει των συναδέλφων εξ των πολιτικών τους ομάδων και ακολουθούν τώρα οι ατομικέ τοποθετήσεις. Οι προσωπικές. Για δύο λεπτά πρώτος ο κύριος Μπαλντασάρη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Θα ψηφίσουμε αύριο την έκθεση Ζάιερ και θα, θα ψηφίσουμε ουσιαστικά για ένα νέο μέσο το οποίο προβλέπεται συνθήκη τη Λισαβόνα, τι εκτελεστικέ πράξει και τι κατεξοδότηση πράξει που αντικαθιστούν ουσιαστικά το σύστημα τη επιτροπολογία. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την έγκριση των πράξεων, θα υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχο από τα κράτη-μέλη όσον αφορά τι εκτελεστικέ αρμοδιότητε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικός ο κανονισμός αυτός και έχει πολύ μεγάλη σημασία και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τη Διοργανική Συμφωνία. Χάρη στην καλή συμμετοχή, έστω και καθυστερημένη, όλων των επιτροπών, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε σε πρώτη ανάγνωση την, τον κανονισμό αυτό, την πρόταση κανονισμού. Πιστεύω ότι θα μας επιτρέψει το νέο αυτό σύστημα να καλύψουμε τις προτεραιότητες της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ότι θα καταφέρουμε ουσιαστικά να έχουμε ένα καλύτερο έλεγχο εξ ονόματος του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δημιουργηθεί μια επιτροπή προσφυγής που θα προεδρεύει αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καταφέρουμε να έχουμε και μια ρήτρα αναθεώρησης που θα μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας. Εν κατακλείδη θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα εμπόδιο το οποίο είχαμε. Το πώς θα καταφέρουμε να συμπεριληφθεί η κοινή εμπορική πολιτική στον κανονισμό αυτό. Μολονότι η τελική συμφωνία επιτρέπει σε μια μεταβατική περίοδο 18 μηνών να χρησιμοποιηθεί η απλή πλειοψηφία για την έγκριση των πράξεων anti-dumping, στη συνέχεια τα μέτρα αυτά θα υπαχθούν στο σύστημα της ε, ενισχυμένης ε, πλειοψηφίας, της ειδικής πλειοψηφίας. Ήταν πολύ δύσκολο να πετύχουμε τη δύσκολη αυτή συμβαστική λύση και ελπίζω ότι αυτό θα βρει σύμφωνου τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση και του ηθήνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τον ίδιο τον εμπορικό κλάδο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίο ο ο κύριο Σούστα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν συμφωνώ με του ε, προελίσσαντε, του τελευταίου τουλάχιστον που μίλησαν. Θεωρώ ότι ε, όλη αυτή η πρόταση που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν σέβεται το πνεύμα της συνθήκης Λισαβόνας. Ουσιαστικά θέλουμε αυτή τη στιγμή ένα 70% των προτάσεων να περνάνε σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο και δεν πιστεύω ότι θα πρέπει σε πρώτη ανάγνωση να κλείσει ε, ένα τέτοιο νομοθέτημα το οποίο έχει να κάνει με την ίδια την ισχύ και τις αρμοδιότητές μας στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις πράξεις anti-dumping. Θεωρώ ότι εδώ πέρα περνάμε από ένα καθεστώς ασφάλειας δικαίου σε πρωτοβουλία των κρατών μελών που ε, ενδεχομένως να οδηγήσει και σε μια αντιπαράθεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Επίσης, αυτή η ρήτρα που προβλέπεται για την ε, αυτόματη προσαρμογή όσον αφορά την ε, πολιτική γεωργίας, θεωρώ ότι αντιβαίνει στις προτεραιότητες και στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε τόσο γρήγορα και βιαστικά σε πρώτη ανάγνωση να καταλήξουμε συμφωνία για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ κύριε Σούστα. Το λόγο τώρα έχει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος Σεύκοβιτς, για να απαντήσει. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σχόλια που ακριβώς δείχνουν πόσο περίπλογο είναι το ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα από τα σχόλια σε σχέση με την αναθεώρηση και τη δέσμευσή μας ε, να το κάνουμε σε όλες τις απαραίτητες πράξεις. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Λένε στο, πλαίσιο της συμφωνίας πλαίσιο. 299 Συν 153 πράξεις πρέπει να ευθυγραμμιστούν και αν θέλουμε να το κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας είναι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Και εντάξει, είπα είναι φιλοδοξία μας, αλλά δεν εννοούσα τη επιτροπή μόνο, εννοούσα όλων των θεσμικών οργάνων, γιατί ακριβώς χρειάζεται τη συνεργασία όλων. Και θα ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο Μίτσελ, έχω το, τρέφω το μέγιστο σεβασμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω, ε, στη δήλωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μία μικρή παράγραφο που λέει τα εξή. Ενώ η διαδικασία αυτή τη ευθυγράμμιση έχει δρομολογηθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα, ε, για τις, ε, για τα, εφαρμοστικά, για τα εκτελεστικά μέτρα τα οποία στο μέλλον μπορεί να γίνουν εκτελεστικέ πράξει. Οπότε η δέσμευσή μα για το μέλλον είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη σε σχέση με την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, θα ενημερώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει όλες τις πληροφορίες ε, όπως και οι επιτροπές. Οπότε ε, έχουμε την πρόθεση να ενημερώνουμε συνεχώς το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λένε γιατί διευκρίνησε την κατάσταση ε, σε σχέση με το ότι αυτό που συζητούμε σήμερα είναι οι εκτελεστικές πράξεις και αυτό δεν προκαταβάλει επουδενή το κατά πόσο θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε κατεξουσιοδότηση πράξης ή εκτελεκτικές πράξεις στο μέλλον. Ε, σε σχέση με το ζήτημα της ευθυγράμμισης, νομίζω ότι ο κύριος Ντεκάστρο δεν ήταν εδώ όταν ε, διάβασα την ε, δήλωση της Βελγικής Προεδρίας και την πλήρη αποσίωσή της ε, στο στόχο της πλήρους ευθυγράμμισης κατά τα ερχόμενα έτη. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι μόνο συμφέρον του Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Βουλίου να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα και θα τιμήσουμε τη συμφωνία αυτή. Όσον αφορά το θέμα του αντι-dumping, ε, ε, ποιο είναι το σύστημα σήμερα Υπάρχει απλή πλειοψηφία των κρατών μελών που σημαίνει ότι κάποιος αντιπρόσωπος μπορεί να μπλοκάρει την, την ε, ε, απόφαση αλλά αυτό χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για να γίνει. Αυτό που λέμε ουσιαστικά είναι ότι ενισχύουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στον ε, τριμερή διάλογο, όπως ακριβώς είχε προβλέψει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω, ε, κύριε Πρόεδρε, τονίζοντας τη σημασία της ασφάλειας δικαίου στην όλη διαδικασία. Γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με ευαίσθητα ζητήματα, όπως το εμπόριο, όπως τα μέτρα αντι-dumping, όπως τα μέτρα... Procedures Πρέπει να έχουμε μια σαφή κατανομή ρόλων και ευθυνών ε, και πρέπει να έχουν τα κράτη-μέλη πολύ συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου που του τα δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας και χρειαζόμαστε ασφάλεια δικαίου για να μπορούμε να κινηθούμε σε αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό νομοθετικό χώρο. Γιατί γνωρίζετε ότι πολύ συχνά τα μέτρα αυτά ε, είναι αντικείμενο αμφισβήτηση σε διάφορα διεθνή φόρα. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν την πρόταση κανονισμού γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τη θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παγκόσμια δρόμενα. Ευχαριστώ. Κύριε Σεύκοβιτς, τελευταίος ομιλητής, ο εισηγητής μας ε, που θα κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για ε, τη συμβολή σας, όχι μόνο σήμερα αλλά και τους τελευταίους εννέα μήνες όσο εργαζόμαστε επί του θέματος αυτού. Πρώτον, ένα διαδικαστικό ζήτημα. Πολλοί συνάδελφοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το γεγονό ότι βιαζόμαστε σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Υπάρχει πίεση από πλευρά του Συμβουλίου. Ε, κοιτάξτε, ε, δεν ε, μπορώ να πω ε, ότι η πίεση ε, ήταν η αντίστροφη. Δηλαδή, εμείς είπαμε στο Συμβούλιο ότι αν δεν, υπάρχει πρώτη, αν δεν υπάρχει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε να καταρρεύσει ολόκληρη προσπάθεια. Όχι, υπάρχει σαφής διεσμευσή και από τα άλλα δύο όργανα. Γιατί όπως και το Κοινοβούλιο, και το είπε και όλας ο κύριος Σεύκοβιτς, υπάρχει θέμα σταθερότητας της συνθήκης της Λισαβόνας όσο αργούμε να εγκρίνουμε τέτοιου είδους νομοθεσία, τόσο θα συνεχίσει να ισχύει η διαδικασία επιτροπολογίας που δεν μας αρέσει γιατί μας δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δεν είναι και λίγο χρονικό διάστημα, εννέα μήνες είναι. Ε, θα μπορούσαμε όντω να κάνουμε δύο αναγνώσεις με πλήρη διαφάνεια και πολλοί συνάδελφοι μπορούν να το πούν αυτό. Ε, ε, είχα συνεδριάσει σε με τους συντονιστές, με σκιώδεις εισηγητές όλων των επιτροπών, ε, με τους προέδρους των επιτροπών ε, και πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνία γιατί ό,τι θέλαμε το πήραμε παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορεί να μην συμφωνούν. Ό,τι μου ζήτησαν οι διάφορε επιτροπέ υπάρχει στο κείμενο. σω όχι με τη μορφή που μου το ζήτησαν. Ο κύριο Δεκάστρο έχει δίκιο ότι το αίτημά του δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει στο συγκεκριμένη έκθεση για τον κανονισμό, αλλά αφορά συγκεκριμένα τι εκταλαστικέ πράξει. Υπάρχει όμω στο πλαίσιο τη δέσμευση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και την προηγούμενη ευθυγράμμιση και το προηγούμενο όμνιμπους και υπήρχε η ίδια δέσμευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπή και τίμησε ε, την δέσμευσή της αυτή με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οπότε πιστεύω ότι μπορώ να εμπιστευτώ τη δέσμευση αυτή και αν δεν τη τηρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ θα υψώσω το ανάστημά μου, όπως κάνει και ο κύριο Δεκάστρο. Από αυτή την έννοια δεν υπάρχει πίεση. Η πίεση προερχόταν από μένα και με καλή συνεργασία σε δύσκολες διαπραγματεύσεις καταλήξαμε σε κάτι το οποίο εγώ πιστεύω ότι ε, μπορεί να βρει σύμφωνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Λυπάμαι για το γενικό κοινό, ε, για το βίτερο κοινό που δεν καταλαβαίνει τη δουλειά που κάνουμε εδώ, αλλά είναι γεγονός ότι η διαφάνεια και ο κοινοβουλευτικό έλεγχο των ζητημάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ καλύτερο μετά από τον κανονισμό αυτό, μετά την έγκριση του κανονισμού αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σάιερ. Όταν μιλάτε για το ευρύ κοινό, ε, αναφέρεστε στον πρόεδρο φαντάζομαι, γιατί δεν έχουμε περισσότερο κοινό αυτή τη στιγμή. Και οι υπόλοιποι είστε υπερηδικοί